κατάσταση αυτή στη Λευκορωσία και θα προτείνει ε, να δοθεί συνέχεια στο ψήφισμα που εγκρίνατε τον Ιούνιο εδώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάλστρομ. Έτσι λίγη συζήτηση για την Λευκορωσία και θα ψηφίσουμε αμέσω μόλις έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για δύο ακόμα περιπτώσεις, η πρώτη από τις οποίες είναι το Σουδάν, η κατάσταση στο νότιο Κορδοφάν και τον γαλάζιο Νείλο. Δίνω το λόγο ευθύ αμέσως για να ξεκινήσει η συζήτηση στον κύριο Τάνοκ. Um, Παρά την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν, παραμένουν κάποιες εντάσεις ε, ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο με την πολιτεία του Γαλάζιου Νείλου και το Κορδοφάν και την περιοχή του Άρμπιγε. Εκεί όλος περιέργως υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και μεγάλες ποσότητες νερού. Εκεί λοιπόν ε, συνάπτονται διάφορες ε, συμμαχίες ανάμεσα στην ε, Χαρτούμ και τις πολιτείες. Η συμφωνία έδωσε πρόβλεψη για δημοψήφισμα στον Γαλάζιο Νείλο και στο Νότιο Κορδοφάνο, ώστε να αποφασίσουν για το μέλλον τους οι πολίτες των περιοχών αυτών. Δυστυχώς ακυρώθηκε το δημοψήφισμα και έτσι υπήρξαν συγκρούσεις ανάμεσα στο Σουδανικό Χαρχό, τον SAF και το SPLA, τον ε, Λαϊκό Μέτωπο Ανεξαρτησίας. Η κατάσταση στο Νότιο Κορδοφάν και στο Γαλάζιο Νείλο επιδεινώνεται ανησυχητικά τις τελευταίες εβδομάδες και φαίνεται να, στόχος να είναι η εθνοτική φυλή των Νούμπα. Έχει υπάρξει εισβολή του Σουδανικού στρατού στο Νότιο Κορδοφάν και στο Γαλάζιο Νείλο. Ο εγκληματίας πολέμου Μπασίρ και το καθεστώ του θα πρέπει μονομερώς να δηλώσουν πάυση του πυρός για να μην υπάρξει επιπλέον αιματοχυσία. Η Χαρτούμ επίσης θα πρέπει να τηρήσει τις νομικές της υποχρεώσεις ε, προσκολώντας και τηρώντας τις συμφωνίες που υπέγραψε το 2005. Είπα τους εκπρόσωπους μαζί με τον ε, Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ έχουν καταδικάσει τον ε, την κλιμάκωση της βίας γιατί αυτές οι συγκρούσεις μπορεί να ακυρώσουν όλη την καλή εργασία των, ε, της διεθνούς κοινότητας και να επιστρέψουμε στον πόλεμο μεταξύ Βορρά και Νότου. Σας ευχαριστούμε κύριο, κύριε Τάνοκο, ο κύριος Ταβάρες έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Το, Σουδάν, το Νότιο Σουδάν δήλωσε την ανεξαρτησία του, διακήρυξε την ανεξαρτησία του πριν από κάποιους μήνες. Η γέννηση μιας νέας χώρας είναι υπόδεινη και πολύ καλά τα περιέγραψε ο συνάδελφος ε, Τάνο και υπάρχουν εντάσεις στα σύνορα και η σύγκρουση που συνεχίζεται με το Βόρειο Σουδάν. Συνεχίζεται στον Γαλάζιο Νείλο, στον Νότιο Κορδοφάν και έχουμε παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δυστυχώς μας έχει συνηθίσει σε αυτές όμως το καθεστώς του Μπασίρ. Είναι μια από τις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου με πολύ κακές συνθήκες υγείας, μεγάλη θνησιμότητα και φαίνεται να προχωρά σταθερά προς τον πόλεμο με τους βόρειους γείτονές του. Είναι μια χώρα που μόλις γεννήθηκε Μόλις ε, οι Νότιοι Σουδανοί γιόρτασαν την ανεξαρτησία τους και ήδη αισθάνονται πως δεν έχουν χώρα γιατί η γη εκεί κοστίζει τρία λεπτά το εκτάριο. Οι ξένες εταιρείε αγοράζουν εκατομμύρια εκταρίων στην Νότια Σουδάν για να έχουν πρόσβαση στις υπόγειους πόρους τους, στις φυσικές, στους φυσικούς πόρους του χωρίς ο λαός του Σουδάν να γνωρίζει τίποτα για όλα αυτά γιατί η κυβέρνηση ασχολείται με τον μεγαλύτερο του γείτονα στην στη σύγκρουση με το Βόρειο Σουδάν, ετοιμάζεται για πόλεμο και δεν δίνει αρκετή προσοχή στις, στο ίδιο την επικράτεια και στους πόρους του. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάμε τέτοιου είδους θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές φορές έχουμε μια θέση η οποία είναι αντιδραστική, ε, ε ε, αντιδρούμε όταν ήδη γίνονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν έχουμε μια συνεχή εικόνα, δεν δίνουμε προσοχή όταν, γίν, όταν συμβαίνουν οι παραβιάσεις και δεν δίνουμε σημασία σε αυτό του είδους της, ε, την ανεξαρτησία ακριβώς τη στιγμή που μια χώρα είναι νέα, είναι ευάλωτη και πρέπει να προστατεύεται με συγκεκριμένο τρόπο, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και απ' έξω ε, δέχονται επιθέσεις οι ευρωπαϊκές εταιρείες, κινέζικες εταιρείες, ε, αμερικανικές εταιρείες που αγοράζουν την ε, γη μεταμανίας. Δεν θα υπάρχει μέλλον για αυτή τη χώρα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτό το λέω στον μόνιμο εκπροσωπό μας στο Νότιο Σουδάν, ώστε να κάνει προσπάθεια στη δικό μας εικόνα και η συνοδεία σε αυτή τη χώρα να είναι συστηματική και συνεχής και όχι μόνο κατά κατά περίπτωση όπως γίνεται τώρα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βερζιά είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, το δημοψήφισμα για αυτοδιάθεση και η πρόσβαση στην ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν ε, μας οδηγούσε να ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μία ειρήνευση, πράγμα όμως το οποίο δεν προχώρησε όσο δεν λυθεί το θέμα των συνόρων μεταξύ των δύο κρατών λόγω της οικονομικής και στρατηγικής σημασίας αυτής της πετρελαιοφόρας περιοχής. Και το, οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι πλήττονται ιδίω από σκανδαλώδεις αεροπορικές επιθέσεις και διότι η μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν μπορούν να παρέμβουν διότι αυτοί οι οποίοι τροφοδοτούν με ε, όπλα τους ε, ε, εμπόλεμου ε, είναι τη μία η Κίνα και η Ρωσία και την άλλη οι Ηνωμένε Πολιτείε. ενώ θα μπορούσαν να διευκολύνουν το έργο των προσώπων του ΟΗΕ και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μία βελτίωση της καταστάσεως η οποία θα υλοποιηθεί. Η κυρία Ντεκάιζερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το ψήφισμα είναι πολύ πολιτικό όντως διότι αυτό το οποίο κρύβεται πίσω από ε, τις εξάρτησεις και την τωρινή διαμάχη είναι αυτά τα οποία δεν ελήθησαν ε, ε, στην συμφωνία της ειρηνευτικής διασκέψεως του 2005. Οπότε είχε λεχθεί ότι προτού προχωρήσει στην ανεξαρτησία το Νότιο Σουδάν έπρεπε να, γίνει, να γίνουν ελεύθερες εκλογές που έγιναν ότι έπρεπε έπρεπε να υπάρξει ένα δημοψήφισμα αλλά και πριν από όλα αυτά πολλά άλλα προβλήματα έπρεπε να έχουν λυθεί. Και δεν μιλώ για τον καταμερισμό του πετρελαίου, ε, των δικαιώματων ε, των νοτίων που ε, είχαν δικαιώματα στο βορρά, το θέματα το θέμα το, της ηθαγενείας αλλά τόσα πολλά αλλά μείνανε σε εκκρεμότητα διότι δεν υπήρξε συμφωνία. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά εάν δεν γίνει καταρχήν το δημοψήφισμα, δεύτερον να γίνουν οι δύο διαβουλεύσεις και στον Μπλε Νίλο και στο Νότιο Κορδοβάν και να μπορέσει η διεθνής κοινότης να επέμβει για να λύσει το πρόβλημα. Οι στρατευμένοι είναι ανεξέλεγκτη και ιδίως αυτή του, ο στρατός του Νοτιού Σουδάν που δεν είναι καλά οργανωμένος και γι' αυτό ζητήσαμε το ICC να εφαρμοστεί και ο Μπασίρ να προσταχθεί στο δικαστήριο της Χάγης. Αλλά εδώ μιλάμε για πολιτική απόφαση ε, θεμάτων που έχουν μείνει ατελεί. Η κυρία Όγιουλαντ. Πρόεδρε, η σύγκρουση στο νότιο Κορδοφάν και στο γαλάζιο Νείλο έχει οδηγήσει στην εκτόπιση 200.000 ατόμων σύμφωνα με εκτιμήσεις. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας του γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν παίρνουν την άδεια για να δουλέψουν επί τόπου. Πρέπει να επενθυμίσω ότι κατά το δεύτερο φίλιο πόλεμο στο Σουδάν 1983 δηλαδή με 2005, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, οι περισσότεροι απλοί πολίτες, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ε, λοιμού. Επαναλαμβάνεται τώρα μια τέτοια ανθρωπιστική κρίση, πολύ φοβάμαι. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποφύγουμε. Γι' αυτό και να κάνουμε έκκληση για πάυση, κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσει διαπραγμάτευση για να βρεθεί μια πολιτική λύση στη σύγκρουση και να επιτραπεί στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να πάνε και να βοηθήσουν τον κόσμο και στο Νότιο Κορτοφάν και στον Γαλάζιο Νείλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως μπορούν όλοι να δουν, σπάνια έχουμε καλά νέα από το Σουδάν. Και γι' αυτό ακριβώς ξανά και ξανά μιλάμε για το θέμα αυτό. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε την ανεξαρτησία του Νότιου Σουδάν. Κάτι το οποίο επισκιάστηκε από τις συγκρούσεις τις βίες συγκρούσεις στο νότιο Κορδοφάν του Ιουνίου. Αυτό εννοώ τώρα. Και μόλις υπεγράφει συμφωνία το Σεπτέμβριο για την περιοχή Αμπέι, ξέσπασε νέες βιαιότητες στο νότιο Κορδοφάν και στο γαλάζιο Νείλο. Γι' αυτό και η κατάσταση θυμίζει σαν να πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Και γι' αυτό ακριβώς όλες οι αρχές της περιοχής δεν έχουν πια αξιοπιστία. Συμφωνώ με τους συναδέρφους και κάνω και εγώ έκκληση στον πρόεδρο Μπασίρ να σταματήσει αυτή την κατάσταση και πιστεύω και εγώ όπως και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να καταλήξει στο δικαστήριο. Η συμφωνία της βέβαια πάντως τον Ιούνιο και είναι κάτι που θέλει να αποκλειστεί η στρατιωτική λύση. Και γι' αυτό και με εκπλήσει το γεγονός ότι το Σουδανικό Κοινοβούλιο τάθηκε υπέρ της στρατιωτικής λύσης. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ακριβώ πρέπει να αποφύγουμε. Η κυρία Σάγια έχει τώρα το λόγο που μιλάει εκ μέρους του ΕΛΚ.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 μη κυβερνητικές οργανώσεις λέγουν ότι χιλιάδες πρόσφυγες έχουν φύγει από την Αιθιοπία και ο στρατός λέγει ότι σε μία περιοχή υπάρχουν ακόμη ένοπλες σειράξεις. Αποδεικνύεται ότι περίπου 20.000 μέτρα έχουν φτάσει στην Αιθιοπία φεύγοντας από τον πόλεμο και οι διεθνείς οργανώσεις ε, έχουν ζητήσει από το Σουδάν να σταματήσει ε, να βομβαρδίζει τον νότιο Κορδοβάν το οποίο βομβαρδίζει συνεχώς και έχει επίσης λεχθεί ότι αυτές οι επιθέσεις κατά των πολιτών μπορούν να θεωρηθούν και ε, ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος ζητάτε να αναλάβουμε μέτρα και αν αυτό δεν είναι δυνατόν θα έπρεπε ε, διεθνώς να γίνει μια τέτοια οργα ανάλυση καταστάσεως. Η ε, κυρία Γκόμες, έχοντας παρακολουθήσει το τι έχει συμβεί και επειδή έχω επισκεφθεί την Ζούμπα πριν από το δημοψήφισμα για την εξαρτησία, λυπούμε, αλλά δεν με εκπλήσει η κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα του Βορείου Σουδάν και των Νοτιών Πολιτιών. Αυτοί που είναι στη διεθνή κοινότητα, δηλαδή η ΕΠΑ, η Αφρικανική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εθελοτυφλούν απέναντι στις εγκληματικέ ενέργειες του Προέδρου Μπασί, συμβάλλουν στην ατιμορρησία του γιατί δεν τον αναγκάζουν να πάει στην Χάγη. Θα πρέπει να δεχτούμε όλοι κάποια ευθύνε για αυτή τι εξελίξει όπου χάνονται ανθρώπινε ζωέ και ε, δεν επιτρέπεται καν η πρόσβαση στι ανθρωπιστικέ ε, οργανώσει. Τα περισσότερα από όσα συστήνει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι λογικά. Αλλά πραγματικά αμφιβάλλω, θα σα το πω, ε, για το κατά πόσο θα υπάρξει πρόοδος στην επίλυση της ε, σύγκρουσης που είπε η συνάδελφος Βερονίκη Τεκεζέρη είναι πολιτικής φύσης ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο εάν εξακολουθήσουμε δηλαδή να ε, θέτουμε τις ε, ελπίδες μας σε τέτοιους ανθρώπους όπως ο κύριος Στάμπο Μπέκη πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ο κύριος Πάσκα. Κύριε Πρόεδρε, Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι εδώ και ο καιρό λέγουν ότι παρακολουθούν τον κύριο Μπασίρ αλλά δεν πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να ισχύσουν δύο, δύο κράτη σε αυτή την περιοχή. Η διαγραφή των συνόρων ε, ακόμη ε, εκρεμεί και τα τελευταία γεγονότα στο νότιο ο Κορδοφάν ε, αποδεικνύουν ότι παίζει κανείς με την φωτιά και ε, ε, έτσι κινείται ο πρόεδρος ενώ η μοίρα των ανθρώπων η οποία κινδυνεύει τον αφήνει τελείως αδιάφορο και υπάρχουν φυλακισμοί όλων αυτών που δεν του δεν πρόσκυνται στον ε, πρόεδρο γι' αυτό και θα πρέπει μαζί με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις Ηνωμένε Πολιτείε να προσπαθήσουμε να εξασκήσουμε διπλωματική και οικονομική πίεση στον Ελμπασίρ για να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του να βοηθήσουμε το λαό του Κορδοφάν για να του επιτρέψουμε μία ε, αξιοπρεπή διαβίωση. Ο κύριος ε, Όμπερ Μάγερ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου ε, ε, ε, η κυβέρνηση της, του Σουδάν έχει ανακοινώσει η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με ε, σειράξεις και με πολλές διαφυγές ατόμων μέσω, προς την Αιθιοπία. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με το Διεθνές Δικαστήριο των ε, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητος και να μπορέσει να σταματήσει η ατιμορρησία εις το Σουδάν και ε, να ε, ξεκινήσει η ε, δίκη του κυρίου Ελμπασίρ για να μπορέσει να υπάρξει ένα κράτος δικαίως διότι διαφορετικά υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρξουν αποτυχημένα κράτη failed states σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Ομπερμάγερ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ. Η κυβέρνηση του Σουδάν κάνει δολοφονίες, αλλά εμποδίζει τον υπόλοιπο κόσμο να ανακαλύψει την αλήθεια. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν πρέπει να συνεχίζει να κοιτάει από την άλλη πλευρά, αλλά να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Εμείς τουλάχιστον εδώ σήμερα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τον Ιούλιο έγινε ανεξάρτητο το Νότιο Σουδάν. Δυστυχώς όμως δεν ακολούθησε ειρήνη το γεγονός αυτό. Πολύ το διαπιστώνουμε και το έχουμε ακούσει από παλιά από ένα γνωστό Σουδανό που είδε από το 1981 έλεγε ότι η χώρα μου υποφέρει και θα υποφέρει πάντα. Η χώρα είναι πολύ πλούσια, αλλά δεν μπορεί να αποφεληθεί τους πόρους της. Πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να φτάσει η ειρήνη στην περιοχή και να μπορεί ο κόσμος να αποφεληθεί από τις σοδιές του και να ζήσει σε ειρήνη. Ευχαριστούμε. Κυρία Φενισίνη, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, στα πλαίσια του ψηφίσματος αυτού υπάρχουν δύο πτυχές πολύ σημαντικές. Απ' τη μια είναι η προστασία του πληθυσμού, των πολιτών από τους βομβαρδισμούς. Εξαιτία των βομβαρδισμών αυτών, ο κόσμος αναγκάζεται να φύγει από τα σπίτια του, ζει κάτω από φρικτές συνθήκες, χωρίς να έχει τι να φάει. Πρόκειται για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο πρέπει να σταματήσουμε. Το Νότιο Κορδοφάν επιγόντω χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια από πλευράς ε, άλλων χωρών, από πλευράς επίσης μη κυβερνητικών οργανώσεων και πρέπει να υπάρξει διάλογος ώστε να φτάσουν τρόφιμα στην περιοχή. 200.000 άνθρωποι, εκ των οποίων 70.000 γυναικόπαιδα, χρειάζονται επιγόντως τη βοήθεια αυτή. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να φτάσει εκεί η βοήθεια και πρέπει να φροντίσουμε να φτάσουν και παρατηρητές, ανεξάρτητοι παρατηρητές παρακαλώ, για να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή. Ε, ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, κύριε ο κύριος Ντες, εδώ και πολλά χρόνια μιλάμε στο Κοινοβούλιο για την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν, όπου υπάρχει ουσιαστικά ένας κατά πλειοψηφία ε, χριστιανικός πληθυσμός, ο οποίος υποφέρει ε, πάρα πολύ και οι δυνάμεις του Προέδρου Αλ Μπασίρ ουσιαστικώς έχουν προβεί σε μία γενοκτονία με βιασμούς, με απελάσεις γι' αυτό και δεν κατάλαβα αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ερντογκάν προσβάτος ο οποίος είπε ότι εν αντιθέσει με την λωρίδα της Γάζας δεν διαπιστώ διαπιστώνει γενοκτονία στο Νότιο Σουδάν και μια τέτοια χώρα θέλει να προσχωρήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς σαν Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε το λαό του Νοτιού Σουδάν και να είμαστε ανοιχτοί κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να τους εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία για τις συγκρούσεις στο νότιο Κορτοφάν και στο Γαλάζιο Νείλο που ξέσπασαν την 1η Σεπτεμβρίου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν και τις δυνάμεις του Σεδικού Σουδανικού Λαϊκού Κινήματος Απελευθέρωσης. Οι συγκρούσεις αυτές έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα βίες και έχουν σαν αποτέλεσμα να χαθούν πάρα πολλές αθώες ζωές και να εκτοπιστούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει εξάπλωση όμως της ε, βίας και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται επιγόντως βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια για τους ανθρώπους αυτούς. Όσο γίνεται πιο γρήγορα επίσης πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ε, δύο πλευρές. Πρέπει να βρεθεί ένας πολιτικός διακανονισμός, είναι ζωτική σημασία για τη χώρα και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Ως Ευρωβουλευτής κάνω έκκληση και στις δύο πλευρές να πάψουν τις εχθροπραξίες και να σταματήσουν κάθε πράξη βίας. Και επιπλέον ζητάω και στις δύο πλευρές και στη διεθνή κοινότητα να πάρουν ό,τι μέτρα χρειάζεται για να διασφαλίσουν την προστασία όλων των Σουδανών πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κρετού είναι η επόμενη. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, δυστυχώς η γέννηση μιας νέας χώρας την 1η Σεπτεμβρίου δεν οδήγησε και στην ειρήνη, μια που 200.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή τα σπίτια τους εξαιτίας της κλιμάκωσης της βίας. Δεν έχουμε επίσης πρόσβαση στο νότιο Κορδοφάνη, στο Γαλάζιο Νείλο. Όπως λέει και η έκθεση του Human Rights Watch του Αυγούστου, οι στρατιωτικές δυνάμεις παραβιάζουν κάθε διεθνή συμφωνία και έχουν σαν αποτέλεσμα να είναι θύματα βίας ακόμα και οι υπάλληλοι του ΟΗΕ, επεσταλμένοι του ΟΗΕ εκεί. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίσει ατιμωρητή, ιδιαίτερα που όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν κάλλιστα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πρέπει πρώτα να πάψουν οι εχθροπραξίες και στη συνέχεια να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους πολίτες εκεί. Πρέπει να εφαρμοστούν οι συμφωνίες ε, για την περιοχή Αμπέη που έχει δεχτεί ο πρόεδρος του Νότιου Σουδάν. Αυτό αποτελεί μια ελπίδα εφόσον εμπλεχτεί και η διεθνής κοινότητα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σόνικ. Κύριε Πρόεδρε, κατά διάρκεια αυτής της σύγκρουσης όπου οι επιθέσεις της βόρειας κυβέρνησης γίνονται εναντίον της νότιας κυβέρνησης, θα πρέπει να φροντίσουμε για την τραγική κατάσταση του αοπλού πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση στα τρόφιμα, σε νερό. Η κατάσταση δεν επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι οργανώσεις που θέλουν να βοηθήσουν δεν έχουν πρόσβαση στον πληθυσμό αυτό που αντιμετωπίζει τέτοιε δυσκολίε. Τα αποθέματα που υπάρχουν στη χώρα εξαντλούνται και η διεθνή κοινότητα πρέπει πραγματικά να ενεργήσει, να δραστηριοποιήσει οι πολίτες δεν μπορούν να αμυνθούν ε, κατά των βομβαρδισμών μόνοι τους. Τα υπεύθυνα άτομα για την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης ε, θα έπρεπε να ε, τιμωρηθούν όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέπο αυτή η δημιουργία του νέου κράτους του Νοτιού Σουδάν τον Ιούλιο εφέτος δεν οδήγησε στην ειρήνη διότι διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες ακόμη βομβαρδίζονται και αυτό αποδεικνύει ότι ο πρόεδρος του Σουδάν Ελ Μπασίρ δεν ενδιαφέρεται για να επιλύσει ειρηνικά το θέμα. Υπάρχει όμως, υπάρχουν ανθρωπιστικές δεσμές όταν υπάρχει μία στρατιωτική ε, και ένοπλη σύραξη και θα πρέπει να επέμβει η εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να προωθήσει μία πολιτική λύση της καταστάσεως του Νοτιού Σουδάν. Ευχαριστώ. Και τέλος... Κύριε Πρόεδρε, η διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Νοτιού Σουδάν δεν έλυσε το πρόβλημα αντιθέτων ε, δημιούργησε προβλήματα μεταξύ των πολιτών και υπάρχουν νέες ε, προκλήσεις μπορεί να υπάρξει ε, μια κατάσταση η οποία θα μεταδοθεί και στα άλλα κράτη και ε, δεν επιλύεται η κρίση. Παραμένει όμως και ένα άλλο πρόβλημα, δηλαδή η ανθρωπιστική βοήθεια και η κατάσταση λήψεως τροφίμων έχει οξυνθεί και οι δυνάμεις ασφαλείας στο νότιο Σουδάν έχουν κατηγορηθεί ε, διότι εμποδίζουν την, το ανθρωπιστικό έργο των ε, οργανώσεων. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει μία, ένας διόλογος ε, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν οι ε, οργανώσεις ε, που αναλαμβάνουν τη βοήθεια. Πριν δώσω το λόγο, ο κύριος Πόσελτ, πριν δώσω το λόγο στην Επίτροπο. Δέχεστε την μπλε κάρτα, ο ναι, Συγχωρείτε, ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο αν θεωρεί ε, ότι πρέπει ήδη να θεωρήσουμε αποτυχημένη την προσπάθεια του Νοτιού Σουδάν αντί να το βοηθήσουμε και να το στηρίξουμε. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι από την ομιλία μου μπορούσε κανείς να εκλάβει κάτι τέτοιο, διότι θα ήθελα βεβαίως να δώσουμε μία δυνατότητα στο Νότιο Σουδάν. Επίτροπε, θα δώσουμε μια ευκαιρία στο Νότιο Σουδάν. Φυσικά, Πρόεδρε, νομίζω πως ναι. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που θέσατε στο επίκεντρο της συζήτησης την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν και στον Γαλάζιο Νείλο. Εν γέννη θα πρέπει να δείξουμε ότι ένας πόλεμος χωρίς εικόνες δεν είναι ένας ξεχασμένος πόλεμος. Η κυβέρνηση του Σουδάν περιορίζει την ανθρωπιστική βοήθεια στο νότιο Κορδοβάν και στην πολιτεία του Γαλάζιου Νείλου. 50.000 πολίτες έχουν φύγει από την πολιτεία αυτή και 200.000 έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση στο νότιο Κορδοφάν. Δεν είναι εύκολο να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει επί τόπου για να βοηθήσουμε τους πληθυσμούς που, που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Πριν από λίγες εβδομάδες αποφασίσαμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και ο ΙΕ το ίδιο έκανε και το ίδιο φυσικά ισχύει τώρα για το, την πολιτεία του Γαλάζιου Νείλου. Παρά τους περιορισμούς που είχαμε, κάποια βοήθεια δίνεται, ιδιαίτερα χάρη σε προηγούμενη τοποθέτηση ανα, υλικού σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Ε, στην... Η, ανθρωπιστική βοήθεια είναι 100 εκατομμύρια ευρώ και 40 εκατομμύρια ευρώ από την ε, πήγουσα ε, βοήθεια. Έτσι πιστεύουμε ότι θα διατηρηθούν οι προσπάθειες ανακούφισης και στα δύο Σουδάν, ενώ αυξάνονται οι ανθρωπιστικές ανάγκες στο Νότιο Κορδοφάν και στο Γαλάζιο Στήλ, Νείλο. Ε, βέβαια, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολύ σοβαρέ γίνονται. γίνονται. Υπάρχουν αναφορές για βομβαρδισμούς σε ε, πολιτικούς ε, στόχους, αυθαίρετες ε, κρατήσεις και συλλήψεις και συγκεκριμένες στοχοθετημένες επιθέσεις. Επίσης έχουμε αναφορές για σφαγές και εκτεταμένες λαϊλασίες. Η κατάσταση πραγματικά είναι, χαρακτηρίζεται από δυσανάλογη χρήση βίας και την έλλειψη διάκριση ανάμεσα σε πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους. Πολλοί άνθρωποι γίνονται στόχοι μόνο και μόνο μόνο λόγω της εθνοτικής τους ε, διαφοράς. Ε, ε, συνεχίζονται, συνεχίζεται η βία και καλούμε ωστόσο εμείς τα μέρη να βρουν μια ειρηνική λύση. Η εκπρόσωπη μας στο Σουδάν έχει καλέσει τους διάφορους συνομιλητές σε Χαρτούμ για να περάσει το ίδιο μήνυμα. Επίσης συντονιζόμαστε με την Αφρικανική Ένωση, τον ΟΗΕ και τη ΣΥΠΑ ώστε να εξασφαλίσουμε κοινή προσέγγιση. Στηρίζουμε τις, τις προσπάθειες δια ε, ε, ε, μια μεσολάβηση του Προέδρου Μπέκη. Η ειρηνική συμβίωση είναι προαπαιτούμενο για την συνύπαρξη των δύο Σουδάν, αλλά φυσικά ούτε η σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε συζήτηση για το Σουδάν ολοκληρώθηκε έτσι και θα ψηφίσουμε μετά από την ολοκλήρωση της συζήτησης για το τελευταίο θέμα της σημερινής ημερής διάταξης που είναι η Ερυθρέα και συγκεκριμένα η περίπτωση του